Σας ευχαριστώ. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ο σχετικός κανονισμός ψήφισε αυτή την έκθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να υπόκειται σε αυστηρότερους κανονισμούς. Ως Ουγγαρέζα είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα γιατί ε, γίνονται καταχρηστικές λειτουργίες από πλευράς των ε, τραπεζών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και βλέπουμε στην πράξη του σούγκρους πολίτες που διαμαρτύρονται Παρά τις τραγωδίες που έχουν προκληθεί λόγω των δανείων σε ξένο νόμισμα, οι τράπεζες εξακολουθούν να επιβάλλουν υπηρεσίες και διάφορα προϊόντα στους πολίτες της ε, χώρας μου, στα αεροδρόμια και σε άλλους τομείς. Θα πρέπει λοιπόν, και σε άλλα μέρη μάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να ρυθμιστούν αυτές οι πρακτικές. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mūsdienu ekonomika vairs nav iedomājama bez elektroniskam finansēm. οικονομία σήμερα ε, δεν θα ήταν α, ε, δυνατό να λειτουργήσει χωρίς ηλεκτρονικές συναλλαγές. Παλιά πλήρωνε κανείς ε, χέρι με χέρι. Στη σύγχρονη κοινωνία οι χρηματοοικονομικές ε, ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι λίγο και πιο ε, συχνές, γι' αυτό και θα πρέπει να διέπονται από πολύ ε, συγκεκριμένη νομοθεσία. Γιατί έτσι θα είναι πιο εύκολο να διαχειριστούμε και να ελέγξουμε αυτές τις αλλαγές. Πρέπει να είναι διαφανές το σύστημα ώστε στην αστερική αγορά να μπορούμε να αναπτύξουμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Έτσι θα έχουμε τυποποίηση των συναλλαγών, ε, προμήθεια, των ε, διαμεσολαβητών, όλα αυτά πρέπει να ρυθμιστούν. Είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία της Ένωσης, αλλά και για να έχουν εμπιστοσύνη καταναλωτές. Ε, ο κύριος Πόλτσιακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υποστήριξα την ε, πρόταση του συναδέλφου Ταγιάννη Πιστεύω ότι το να δημιουργηθεί ένας χώρος για τις ηλεκτρονικές αναλλαγές και να προστατεύονται οι καταναλωτές είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό και πολύτιμο. Γι' αυτό και στήριξα την πρόταση αυτή. Το να δημιουργήσουμε έναν ενοποιημένο χώρο για αυτού του είδους τις συναλλαγές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα να εξασφαλίσουμε ένα περιβάλλον ασφαλές. Μιλάμε για την ηλεκτρονική εντολή εμβάσματος ή τις κεφαλαγορές. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά εργαλεία που πρέπει να λειτουργούν ικανοποιητικά και οι συμπολίτε μα πρέπει να ενημερώνονται έτσι ώστε να διευκολύνονται. Ευχαριστώ, Σον Κέλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή. Νομίζω πως ο κύριος ε, Ταγιάννη έκανε σπουδαία δουλειά. Θα ωφεληθεί πολύ ο κόσμος σε αυτό το τομέα, διότι όλα είναι και περισσότεροι συναλλαγές γίνονται διασυνοριακά και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σαφείς κανόνες για όλα αυτά. Στη χώρα μου ε, υπάρχουν πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες φτιάχνονται και θα εξάγουν στο μέλλον ε, αγαθά μέσω ίντερνετ. Οπότε για το λόγο αυτό ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ενδυνάμωση της ενίας αγοράς για να μπορούν να γίνονται σωστά αυτές οι συναλλαγές. Όλα αυτά λοιπόν βοηθάνε πάρα πολύ. Ο κύριος Ποσπισίλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ψήφισα υπέρ της πρότασης αυτής γιατί η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ιδίω των διασυνοριακών ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολύ σημαντική πτυχή ε, για τη δημιουργία της ε, εσωτερική αγοράς. Συζητήσαμε ε, πόσο σημαντική είναι η καλύτερη συνεργασία για τα δικαστικά ζητήματα, πόσο σημαντική είναι η διασύνδεση των αγορών, η εμπορία αγαθών ηλεκτρονικά κτλ. Όλα αυτά τα μέσα θα οδηγήσουν σε κάτι πολύ σημαντικό κατά μένα, δηλαδή στην ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό καλωσορίζω την πρόταση και συμφωνώ με όλα όσα αναφέρονται στη δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών, καταγγελίες και τα λοιπά. Ε, βέβαια, αυξάνεται η επιβάρυνση, μάλλον μειώνονται τα τέλη, όπως τα τραπεζικά τέλη, προστατεύονται καλύτερα τα προσωπικά δεδομένα. Όλα αυτά είναι σημαντικά για τους πολίτες και γι' αυτό θεωρώ σωστή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ε, Όσον αφορά την νομοθεσία για τις ε, υποθήκες και τα ε, χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου στην Ισπανία, η κυρία Μορβάη έχει το λόγο, γιατί η κυρία Κοζάλης απουσιάζει természetesen igennel szavaztam arra a jelentésre amely. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή η οποία έχει ως σκοπό να βοηθήσει όσους έχουν πάρει δάνεια ανυπόθηκα. Θα ήθελα να σας αναφέρω λοιπόν ένα αριθμητικό στοιχείο. Στην Ισπανία υπάρχουν 95 οικογένειες που χάνουν τα σπίτια τους για το λόγο αυτό και στην ε, Ουγγαρία είναι ακόμα πιο δραματική η κατάσταση όπως είπα και στην προηγούμενη παρέμβασή μου Όσοι έχουν πάρει δάνεια σε ξένο συνάλλαγμα δεν θα προστατεύονται πλέον από το μνημόνιο και ο κόσμος θα χάσει τα σπίτια του. Προκειμένου λοιπόν να μπει ένα τέρμα σε αυτή την κατάσταση, οι δικηγόροι και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις θα πρέπει να εξετάσουν την έκθεση αυτή και να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες του. Θα δημοσιεύσω και την έκθεση στην λογαριασμό μου στο Facebook. Ε, Ο κύριος Μάμικινς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ένας από τους βασικούς λόγους που την τελευταία δεκαετία σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και στη δική μου χώρα, ε, ξέσπασε η κρίση, είναι η αδυναμία αποπληρωμής δανείων προς τις τράπεζες για σπίτια, ενυπόθηκα δάνεια και για αυτοκίνητα. Φυσικά θα πρέπει να μπορεί να αποπληρώνει ο ιδιώτης και το δάνειο και τους τόκους, αλλά δεν είναι κανονικός τρόπος αυτός ε, να συνεχίσουν τα πράγματα όταν αδυνατεί τόσος πολύ κόσμος να αποκλειδώσει τα δάνειά τους. Έχει δικαίωμα να έχει κανείς ένα κεραμίδι πάνω στο κεφάλαιο του. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουν τα ρυθμίσεις στις υποθήκες προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να υπερψηφίσει, να ε, αποπληρώνει τα δάνειά του. Ο κύριος Πόλτσακ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα... Ευχαριστώ. Πρέπει να πω δημοσίω ότι δεν υποστηρίζω αυτή την έκθεση. Δεν την υπερψήφισα, γιατί θεωρώ ότι αν τα εθνικά πολιτικά ζητήματα μεταφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα, χωρίς την προσπάθεια εξέβρεσης μιας κοινή ευρωπαϊκής θέσης, δεν υπάρχει πρόβλημα και έχουν χάσει τις, περιουσίες τους τόσες χιλιάδες Ισπανοί λόγω της δραστηριότητας των τραπεζών, τα στεγαστικά αυτά δάνεια και τις υποθήκες. Καταλαβαίνω τι γίνεται και με τις προνομιακές μετοχές κτλ. Ο Πρωθυπουργό της Ισπανίας, η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει κάτι για τα προβλήματα ε, που προέκυψαν επί προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτό δεν μπορώ λοιπόν να δεχθώ. Δεν μπορώ να δεχθώ αυτή την πρόταση. Κυρία Μορβά για το επόμενο θέμα, για τη θανατική ποινή. Είχαμε τη θανατική ποινή μέχρι το 1990 ή 1991, όπως ε, είπε ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο που δίδασκε ποινικό δίκαιο. Εγώ παρακολούθησα δίκες με τους φοιτητές μου όπου επευλήθη η θενοτική ποινή. Τότε εγώ και οι φοιτητέ μου είδαμε ανθρώπους που καταδικάστηκαν σε θάνατο. Επισκεφθήκαμε φυλακές όπου κόσμος περίμενε την εκτέλεση της ποινή του στα ε, κελιά. Από τότε λοιπόν που είδα αυτούς τους ανθρώπους, ε, Βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί είναι πιο δύσκολο για μένα να πω ότι είμαι υπέρ της θανατικής ποινής, ε, όταν ο κόσμος μπορεί όντως να, να θανατωθεί στο δικό μου όνομα, όμως ως, ποινικ, ως δικηγόρος του ποινικού βλέπω φρικιαστικά εγκλήματα που, γίνονται, που διαπράττονται εις βάρος ανθρώπων και παιδιών και γι' αυτό και θεωρώ ότι χρειάζεται η θανατική ποινή. Πώς πισίλ. Πώς πισίλ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 Λύθηκε το πρόβλημα. Okay. Start again. Sorry. Μπορείτε να ξεκινήσετε ε, από την αρχή. Ελπίζουμε ότι λύθηκε το τεχνικό πρόβλημα. No, I, I was Σας παρακαλώ να ξαναπείτε τα, την ε, ομιλία σας γιατί δεν ακούστηκε, δεν μεταφράστηκε μάλλον. Ναι, Πρόεδρε, να επαναλάβω. Εγώ υπερψήφισα αυτή την πρόταση διότι Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω και συζητά, που συζητά διαρκώς τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο θα πρέπει να είναι αυτή που θα αγωνιστεί κατά της θανατικής ποινής. Εξακολουθούν να υπάρχουν 58 Χώρες στον κόσμο που ισχύει η θανατική ποινή και σε ορισμένε χώρε μάλιστα εκτελείται με ιδιαίτερα βάρβαρο τρόπο. Και μιλάω για την Κίνα, την, το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, που είναι χώρε όπου η θανατική ποινή έχει γίνει αντικείμενο κατάχρηση. Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για έναν νεαρό που πρόκειται να εκτελεστεί στη Σαουδική Αραβία σε όλα τα διεθνή φόρα θα πρέπει να προωθήσουμε την κατάργηση της θανατικής ποινής και να επαναλαμβάνουμε πως υπάρχουν εναλλακτικέ ε, στη θανατική ποινή όπως είναι η διαβίου κάθριξη. Ο κύριος Μάμικινς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάθε άνθρωπος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα στη ζωή και σε τρόπους με τους οποίους μπορεί να τιμωρηθεί, ανάλογα με το τι έκανε. Εάν όμως ε, σκοτωθεί, δεν μπορεί να μετανοήσει. Η θανατική ποινή δεν μπορεί να θεωρείται ε, αποτελεσματική στη σύγχρονη κοινωνία. Ε, Ο άνθρωπο δεν μπορεί να χάνει. Και επίσης γίνονται και λάθη. Μπορεί κάποιος να χάσει τη ζωή του, ενώ δεν διέπραξε τελικά το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε πέρσι. Είδαμε να αυξάνονται οι θανατικέ ποινέ, Είναι πραγματικά πολύ λάθο γιατί ιδιαίτερα ε, πολλοί άνθρωποι αποδείχθηκαν τελικά αθώοι. Ε, ο κύριο Κέλλη. Και εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση. Βέβαια είναι ε, ευτυχές γεγονός ότι όλο ένα και περισσότερες χώρες ε, καταργούν τη θανατική ποινή. Είναι εξαιρετικά σημαντικό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην το συζητάμε καν δεν θα έπρεπε τον επαναφορά της θανατικής ποινή. Βεβαίως και διαπράττονται φρικτά εγκλήματα και ο κόσμος εξαγριώνεται και ίσως να θέλει να θανατώσει ή να εκτελέσει κάποιον εγκληματία όμως ο πολιτισμός ε, πρέπει να αναγνωρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ανα πάσα στιγμή. Ε, όπως είπε, επιπόθηκε, πολλοί άνθρωποι έχουν εκτελεστεί και αργότερα αποκαλύφθηκε ότι δεν ήταν οι, οι ένοχοι και γι' αυτό και πιστεύω πως είναι ανθρώπινο δικαίωμα ολόκληρο του κόσμου να μην εκτελούνται οι άνθρωποι. Πρέπει λοιπόν να καταργηθεί η θανατική ποινή. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μακοβέη τώρα. Ευχαριστώ. Είμαι κατά τη θανατική ποινή. Το 2014 θανατώθηκαν 2.500 άνθρωποι ε, λόγω θανατική ποινή. Καθημερινά καταδικάζονται σε θάνατο άνθρωποι για, κοινά, ε, για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου ή γιατί μπορεί να έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους. Παραδείγματος χάρη του διαδηλώνει Και εδώ αναφέρομαι και συγκεκριμένα στην περίπτωση του Αλή Μοχαμέτα Αλ Νίμερο που μας απασχόλησε πιο πριν και ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο λόγω συμμετοχής του σε διαδήλωση. Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία κροτηριάζει τα άκρα, τα, τα μέλη ανθρώπων ε, και για πολύ ε, ε που κάγε καθόλου σοβαρά Τα Πού ζούμε τελικά, το 2015 ζούμε όλοι ή κάποιοι άλλοι όχι. Ευχαριστώ κυρία Σόντροβα. Η κατάργηση της αντικής ποινής ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό ε, και πρέπει να παραμείνει ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι και μια γενική αρχή για τον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. Είναι υψηλότερη αξία άλλωστε η ανθρώπινη ζωή. 2.466 άνθρωποι εκτελέστηκαν το 2014 πιο πολύ στην Κίνα. Στηρίζω το ψήφισμα και το υπερψήφισα όχι γιατί θέλω να εξαγάγουμε τις ευρωπαϊκές αξίες στις άλλες ε, χώρες του κόσμου, αλλά επειδή γίνεται κατάχρηση και εκμετάλλευση της θαντικής ποινή ε, για τις διώξεις πολιτικών ε, αντιφρονούντων ή για άτομα που έχουν διαφορετικό γενετήσιο προσανατολισμό ή διαφορετική θρησκεία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και χαίρομαι που εγκρίθηκε αυτό το κείμενο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, περνάμε τώρα στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την καταστροφή της Ερυθράς ε, Ουγγαρία, η κυρία Μορβάη. Ο στόχος ενός προστίμου ή μιας ποινής είναι η μιας ποινη ειναι Δηλαδή να μην επαναλάβουν το ίδιο αδίκημα στο μέλλον οι ε, δράστες. μετά την καταστροφή της Ερυθράς στην Ουγγαρία. Πρέπει να κοιτάξουμε προς τα εμπρός πια και να εστιάσουμε στην πρόληψη, ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ στο μέλλον κάτι αντίστοιχο. Για να υπάρξει πρόληψη όμως, πρέπει να αντιλούμε ε, διδάγματα και επίσης θα πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες ε, στους δράστες. Γιατί έτσι εξυπηρετείται και ο σκοπός της πρόληψης. Πρόσπιση πριν λοιπόν, πέντε χρόνια η Ουγγαρία επλήγει από μια τεράστια βιομηχανική και φυσική καταστροφή. Πέθαναν δέκα άνθρωποι. 150 τραυματίστηκαν. Συμπάσχω με τις οικογένειες των θυμάτων στην Ουγγαρία. Στην πιο πρόσφατη ιστορία της Ευρώπης είχαμε διάφορες τέτοιες ε, φυσικές καταστροφές. Όπως το 2002 στη Γαλλικία με την πετρελοκυλίδα. Ευτυχώς ε, δεν πέθανε κανείς εκεί, αλλά ε, δεν μπορεί καν να φανταστεί ακόμη ο νους μας ε, τι ε, φυσική καταστροφή συνετελέστηκε. Και βέβαια, δυστυχώς όλα αυτά προήλθαν από ανθρώπινες αυλεψίες. όπως και πολλά βέβαια έχουν να κάνουν τους κανόνες για την αποθήκευση υλικών. Σίγουρα πρέπει να ενημερώνονται όσοι ζουν κοντά σε τέτοιες περιοχές κινδύνου. Ευχαριστώ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 η μεγαλύτερη βιομηχανική καταστροφή που χτύπησε τη χώρα μας, ε, την καταστροφή της κόκκινης λάσπης, ε, τότε υποβάλαμε μια συγκεκριμένη ερώτηση στην Επιτροπή. Πώς θα αλλάξετε την νομοθεσία για να προλάβετε τέτοιου είδους καταστροφές. Πώς θα χορηγήσετε χρήματα ώστε να αντιμετωπιστεί η οικονομική ζημιά που προκλήθηκε από την καταστροφή. Η Κομισιόν δεν απάντησε ποτέ σε αυτές τις ερωτήσεις και γι' αυτό και είμαι δυστυχής που τώρα έχουμε ένα ψήφισμα ε, που υποστηρίζει την αρχή του «Ο Ριπένον πληρώνει» και δεν ε, έχουν καλυφθεί ακόμα οι ζημιές από αυτήν την καταστροφή. Κύριε Μακοβέλη, λείπει, οπότε ο κύριος Κέλλη. Ε, excuse me. We, we now discuss... Α, όχι, συγγνώμη. Τώρα ε, συζητάμε την ε, ισότητα των φύλων. Η κυρία Μορβάη έχει πρώτο το λόγο. Σας ευχαριστώ. Το βασικό νόημα αυτής της έκθεσης είναι ότι χορηγεί χρήματα στις αναπτυσσόμενες, χορηγούνται χρήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι πρόθυμες να λάβουν υπόψη τις ιδέες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτή την αρχή γιατί είμαι κατά των διακρίσεων που βασίζονται στο φύλλο αλλά αυτό που συζητάμε εδώ δεν έχει να κάνει με το δικαίωμα των κοριτσιών να πάνε στο σχολείο στην Αφρική ή με απαγόρευση του ακροτηριασμού των, γεννητικών οργάνων, των γυναικείων γεννητικών οργάνων, γιατί αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο. Λέγεται εδώ στο ψήφισμά μας ότι η ε, άμβλωση είναι ανθρώπινο δικαίωμα και ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει αυτό να το δεχτούν και μιλάμε και για, σε κάποιες παραγράφους για την ε, τα, τους φιλομεταβατικούς και τα λοιπά. Θέλουμε να επιβάλλουμε αυτές τις αρχές σε αυτές τις χώρες με αντάλλαγμα χρήματα και αυτό είναι απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ, Βαμικίνς, η ανθρωπιά Ε, και το ανθρώπινο γένος μάλλον αποτελείται και από γυναίκες και από άνδρες ασφαλώς. Και φυσικά λοιπόν και οι δύο πλευρές αυτές ε, ε, πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι και σε υπερεθνικό επίπεδο θα πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς ακόμα κάποιες γυναίκες κάποιες ηλικία δεν ναι, ελέγχουν απόλυτα τη ζωή τους, ε, εξαναγκάζονται να παντρευτούν, δεν τους επιτρέπεται να πάνε στο σχολείο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να μην υπάρχει καμία διάκριση βάση του φύλου και ασφαλώς και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν ε, πρέπει να υπάρχουν τέτοιε καταστάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρο και η κυρία Μακοβέη δεν είναι εδώ και ο κύριο Κισκέλη λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι ήμουν πολύ ευτυχής που μπόρεσα και εγώ και η ομάδα μου να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης αυτής. Ήταν μεγάλη πλειοψηφία, 520 υπερψήφισαν και αυτό καταδεικνύει ότι κατανοούμε τη σημασία των γυναικών και ότι πραγματικά επιθυμούμε να υπάρχει ισότητα για τις γυναίκες. Αλλά είμαστε και κατά των τροπολογίων 7 και 19 όπου αναφέρθηκε η ελεύθερη διάθεση του δικαιώματος της άμβλωσης στις χώρες αυτές. Δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί τη σωστή προσέγγιση και άρα απορρίψαμε αυτές τις δύο τροπολογίες για το λόγο αυτό. που και δεν εγκρίθηκαν και έτσι καταφέραμε να υπερψηφίσουμε το σύνολο της έκθεσης. Αν ωστόσο η άμβλωση προτείνονταν ευρέως σε διεθνές επίπεδα, θα είχαμε απορρίψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρε και περνάμε στην έκθεση της κυρίας Ζαμπόρσκα και δίνω το λόγο στην κυρία Σόντροβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με την εκθεσία αυτή σε ό,τι αφορά τι ίσε ευκαιρίε και την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στο θέμα εργασία και απασχόληση. Είναι εξαιρετικά ε, σημαντικό το θέμα αυτό και προφανώς το συζητάμε αυτό εκτενώς. Αλλά είναι σημαντικό να το θέτουμε και σε επίπεδο έκθεση. Η κυρία Ζαμπόρσκα έκανε εξαιρετικό έργο και το τονίζω αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλή πρόταση. Και το γεγονός ότι μόνο 364 ε, βουλευτές υπερψήφισαν σημαίνει ότι πολύ απλά δεν ε, καταφέραμε να βρούμε ε, ισχυρή συνένεση. Όλοι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναμείβονται σωστά και ανάλογα με τους άνδρες οι γυναίκες. Είναι όμως κάποιες ε, τροπολογίες και σε κάποιες περιπτώσεις προασπίζουμε την αρχή της επικουρικότητας. Δεν πιστεύω ότι οι ποσοστώσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό αυτό σε ό,τι αφορά δηλαδή τις εταιρείε και το καθεξής. Αυτό ξεπερνά τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου δυστυχώς, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να συλλέξουμε την απαραίτητη υποστήριξη για την πρόταση αυτή που θα αποτελούσε ένα πρακτικό εργαλείο για την ίση αντιμετώπιση και την ίση ανταμοιβή γυναικών και ανδρών. Ακόμα και αν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε τουλάχιστον τα σημαντικά αυτά στοιχεία της έκθεσης που πρότεινε η κυρία Συμπαγόρος. Κύριε Μορβάη. Ε, Ευχαριστώ. Η έκθεση της κυρίας Σαμπόρσκα για τη δεκτική μεταχείριση. Απήχα κατά την ψηφοφορία. Και η ίδια η συντάκτρια της έκθεσης άλλωστε απήχε. Δηλαδή δεν ψήφισε υπέρ της δικής της έκθεσης. Μπορεί για κάποιον που είναι ε, εκτός να μην καταλαβαίνει πολύ καλά, αλλά θέλω να σας εξηγήσω που οφείλεται αυτό. Αξιολογήσαμε και αξιολογούμε συνεχώς το έργο των βουλευτών. Αυτό γίνεται από εξωτερικέ εταιρείε και όλα αυτά γίνονται γνωστά και στον τύπο. Και μπορεί κανείς να πάρει πόντους από το αν έχει κάνει μια ε, καλή έκθεση. Η κυρία Ζαμπόρσκα είναι παγκελματίας Την ανάγκασαν να βάλει ε, τα δικαιώματα για τους φιλομεταβατικούς λοιπά Αλλά αυτό δεν είναι οικείο για αυτήν. Και το κείμενο πλέον δηλαδή δεν μπορούσε να το ε, υπογράψει. Ήταν ευνοχισμένο αν μπορώ να το πω ε, λόγω των τροπολογιών που πέρασαν το κείμενο και δεν μπορούσε να το ψηφίσει ούτε η ίδια η Ορίστε λοιπόν ένα κοινοβούλιο που δεν μπορεί καν να παρεκκλίνει από τις νοσηρές του αξίες και τις ηθικά διαστρεβλωμένες. Η εγγύηση της ισότητας των δύο φίλων, ο κύριος ε, Λινάρ, ε, είναι θεμελιώδης αρχή στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προφανές ότι οι υποψήφοι για μια θέση εργασίας θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλου. Απ' την άλλη πλευρά είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε και ότι οι εργοδότες θα λαμβάνουν υπόψη και θα σέβονται την αναγκαία ιση ευκαιρίες μεταξύ των δύο φίλων. Υπάρχουν βελικέ διαφορές σίγουρα μεταξύ των αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε ε, διακριτική μεταχείριση, γι' αυτό και ψήφισα υπέρ. I voted against this report due to the glaring... Εγώ ψήφισα κατάλληλη, κυρία Σέιμου, λόγω των αντιφάσεων. Στην μία παράγραφο ζητάμε ουδέτερη ταξινόμηση των θέσεων εργασία και στην άλλη ζητάμε δεσμευτική ποσόστοση ε, για τα δύο φύλλα. Ε, και επίση ε, είναι τελείω ακατανόητα ορισμένα πράγματα που γίνονται, που γράφονται. Α αφήσουμε τι γυναίκε και του άντρε να συναγωνίζονται ελεύθερα, χωρί ποσοστό. Σε ελεύθερη κοινωνία ζούμε. Καλύτερα να αφήσουμε έτσι λοιπόν τα πράγματα, να αφήσουμε του ανθρώπου να διεκδικούν τι θέσει με βάση τι τα την αξία τους. Ε, δεν υπάρχει τίποτα θετικό στη θετική διάκριση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκέλη. Σας ξαναευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ε, φανταζόταν κανείς από τον τίτλο ότι όλοι φανεί πέρα αυτής της έκθεσης, όμως πραγματικά κάποιοι έχουμε προβλήματα με μέσα από τις συστάσεις. Αυτό είναι κατανοητό. 344 ε, τελικά από τους 568 ε, συναδέλφους ε, ψήφισαν υπέρ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Εγώ ήμουν υπέρ της έκθεσης με εξαίρεση την τροπολογία 17 και τα τμήματα 1-2 ε, συγκεκριμένα αυτή τη τροπολογία. Το Φιναγκέλ ε, μάλλον καταψήφισε ομαδικά τις τροπολογίε τροπολογίες αυτές, αλλά σίγουρα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να έχουμε ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, στου συντάξους, μισθούς ε, και στις δυνατότητε προαγωγή. Έχουν γίνει αρκετά σίγουρα, αλλά χρειάζεται να ε, θετηθούν οι κανόνες για να έχουμε από εδώ και πέρα και στην ένας πραγματικά ισότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόγκορ. Ευχαριστώ πρόεδρε στην έκθεση αυτή. Δώσαμε μεγάλη έμφαση στην έλλειψη ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ της οικογένειας και της σταδιοδρομίας. Ο το κείμενο επίσης επικεντρώνεται Και το κείμενο αναφέρει λοιπόν και το γεγονός αυτό ως ε, αιτία για την υπογεννητικότητα. Αυτό λοιπόν αποτελεί μια πολύ λυπηρή εξέλιξη για τις κοινωνίες μας και θα καταστεί αυτό ακόμα πιο έντονο φαινόμενο στο μέλλον. Είναι λοιπόν χαρακτηριστική αυτή η απροθυμία τεκνοποίηση ω άμεση συνέπεια τη διακριτική μεταχείριση που υπόκειται οι γυναίκε με μικρά παιδιά. Μιλάμε λοιπόν για την ανισότητα στην άμυβη και αυτό σίγουρα θα μας απασχολήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα το λόγο να δώσω στην εισηγητή την κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πολύ λυπάμαι που δεν κατάφερα τελικά να υπερψηφίσω την ίδια μου την έκθεση και με λυπεί αυτό γιατί η έκθεση αυτή που περιείχε πολλές ε, καλές ε, προτάσεις και συστάσεις. Προσπάθησα να θέσω τα θέματα που προκαλούν διαφορέ μεταξύ ανδρών και γυναικών και τα οποία οξύνονται μετά την απόκτηση του πρώτου παιδιού. Προσπάθησα να τονίσω και άλλε πτυχέ, για παράδειγμα τη ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση γυναικών και ανδρών, όπου και οι γυναίκε ε, τιμωρούνται ουσιαστικά. Αλλά απήχα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας γιατί πέρασαν τροπολογίες με τις οποίες δεν μπορώ να συμφωνήσω και ε, δεν μπορούμε να δεχτούμε κάποια στοιχεία, γιατί αυτό ενδεχομένω να μην οδηγήσει στην ε, ίση αντιμετώπιση και την ίση αμοιβή των γυναικών, γιατί ουσιαστικά φεύγει το στοιχείο αυτό τη γυναίκα που μα απασχολεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τα πρακτικά θα δημοσιευτούν για έγκριση στην αρχή της επόμενης ολομέλειας και αν δεν έχετε αντιρρήσεις θα διαβιβαστούν τα σχετικά ψηφίσματα που ψηφίστηκαν. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση και η συζήτηση.